Κυρίσω την επανεκκίνηση της ε, συνεδρίασης που διακόπησε 8 Οκτωβρίου. Αγαπητοί συνάδελφοι, εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταδικάζω απερίφραστα τις τρομοκρατικές επιθέσει στην Άγκυρα της Τουρκίας. Και εκφράζω στον τουρκικό λαό τη βαθύτατη